Η διάταξη ακολουθεί τώρα η κοινή συζήτηση για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισίας. Η συγκήτρια είναι η κυρία Ντουσαρνέζ. Θέσπιση έκτακτων αυτονόμων εμπορικών μέτρων για την Τινησία και δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισία. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια πρώτα, την κυρία Ντεσάρνεζ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Σεσίλια Μάλμστρομ, κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε ενώπιό μα μια πολύ σημαντική συζήτηση απόψε. Θα επανέλθω σε δύο λεπτά. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου και όλου οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες για το θέμα αυτό, το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για την Τινησία και για την Ευρώπη και για την ιδέα που έχουμε εμείς για την Ευρώπη. Γνωρίζετε όλοι τι γίνεται στην Τινησία. Καταλαβαίνετε όλοι τι δρόμο έχει διανύσει η χώρα αυτή, η Τινησία, από την ε, τελευταία Αραβική Επανάσταση. Είναι από τις μόνες και λίγες χώρες και σπάνιες που κατάφερε τη δημοκρατική μετάβαση και κατάφερε να την εδρεώσει μάλιστα. Άλλωστε, έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και σωστά ε, ο, ο τινησιακός διάλογος και δικαίως. Πάντως γνωρίζετε όλοι και τι προκλήσεις αντιμετωπίζει η χώρα αυτή. Υπήρξαν ε, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, το γνωρίζουμε όλοι, και οι τρομοκράτες δεν χτύπησαν τυχαία την, νησία... αλλά την ε, έπληξαν διότι ακριβώ πετυχαίνει στην προσπάθειά της και ε, ταλαιπώρησαν την οικονομία, δεν υπάρχει τουρισμός, άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, εξαιρετικά υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των νέων πτυχιούχων παρακαλώ, Υπάρχουν όλα τα ζητήματα που τίθεται με την ε, με τη Λιβύη και ίσως αύριο και με την Αλγερία. Βεβαίω λοιπόν θα πρέπει να επιτύχει στην προσπάθειά της η Τινησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τη βοηθήσει να επιτύχει. Αυτό το πνεύμα πριν τα ανέβει στα δύο κείμενα που θα συζητήσουμε απόψε. Το πρώτο κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται για έκτακτα επίγοντα μέτρα υπέρ ε, του ελαιολάδου θα σας εξηγήσω στη συνέχεια περί ως πρόκειται για συγκεκριμένες δράσεις. Όχι απλώς για κούφια λόγια και ωραίες μεγαλεπίπολες δηλώσεις. Θα πρέπει να είμαστε στο ραντεβού της αλληλεγγύης με την Τινησία και τους Τινήσιους. Αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ καλά κάνει είναι όχι να αυξηθούν οι εξαγωγές από την Τινησία, αλλά 35.000 τόνοι επί 2, 70.000 τόνοι, την ποσόστοση ε, χωρίς δεν αυξάνεται λοιπόν η ποσότητα, οι δασμοί. Στην Ευρώπη είναι πάνω από 1.400.000 τόνοι το χρόνο η παραγωγή. Γιατί την τίνηση είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν αποσταθεροποιούν αυτά τα μεγέθη την Ευρώπη. Θα τα ξαναδούμε αυτά του χρόνου, ε, θα τα εκτιμήσουμε και αν υπάρξει πρόβλημα, πράγμα που δεν πιστεύω, σε περίπτωση που υπάρξει θα, θα ληφθούν ε, μέτρα. Δεύτερον, είναι Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Έγινε ένας πρώτος γύρος. Αύριο θα εγκρίνουμε ένα ψήφισμα για το οποίο έχουμε εργαστεί πάρα πολύ στην Επιτροπή μας και το μήνυμα του Κοινοβουλίου είναι απλό. Δεν είναι απλώ ένα ψήφισμα που μιλάει για ελεύθερες συναλλαγές και εμπόριο. Πάνω απ' όλα είναι ένα πολιτικό ψήφισμα που διατρανώνει την υποστήριξή μας και την αλληλεγγύη μας υπέρ της δημοκρατίας, της ανάπτυξης, ε, της οικονομίας στην Τινησία. Λέμε ότι θα πρέπει να είναι πολιτική η συμφωνία, δεύτερο μια συμφωνία ασύμετρη, ασύμετρη. Πρώτα η Τινησία και προοδευτική. Και τρίτον να υπάρξει διαφάνεια. Όχι μόνο διαφάνεια όμως οι Τινήσοι στο σύνολό τους να εστερνιστούν αυτή τη συμφωνία, να την κάνουν κτήμα τους, να την κάνουν δική τους υπόθεση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτό το διάλογο με τους Τινήσιους ε, βουλευτές, τους οποίους υποδεχτήκαμε στο Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εδρεωθούν όλα αυτά με τρόπο μόνιμο και διαρκή. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εξυπηρετεί και την Τινησία και το σύνολο των Τινησίων και τότε και μόνο τότε θα έχουμε έρθει στο ραντεβού των απαιτήσεων των καιρών που είναι να είμαστε παραστάτες στο πλευρό της Τινησίας και των Τινησίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ραπορτέρ. Κυρία Εισηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Σεσίλια Μάλμστρομ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο εξ Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, η Τινησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στενή εταίρια εδώ και χρόνια. Από το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ε, νέα Τινησιακή Δημοκρατία μέσω μιας προνομιακής εταιρική σχέση που δεν περιορίζεται στο εμπόριο αλλά και ε, εκτείνεται και σε διάφορα άλλα θέματα όπως η δυτικοποίηση του πολιτικού διαλόγου και σημαντική αύξηση στην τεχνική και οικονομική βοήθεια προς την Τινησία διότι όπως είπε και η συγγήτρια είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθεί αυτή η χώρα που η δημοκρατία είναι ευάλωτη και αδύναμη και όπου η κατάσταση όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πολύ πολύ δύσκολη για τον τινησιακό λαό και την κυβέρνηση της χώρας. 20 ε, χρόνια μετά από την συνυπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, μετά, ε, μεταξύ μας, όπου το διμερές εμπόριο έχει υπερδιπλασιαστεί, μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία για να βαθύνουμε στις εμπορικές μας σχέσεις ακόμη περισσότερο. Και είναι επιθυσή μου και οι πρόσφατες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες των πολιτών δείχνουν ότι η πολιτική επιτυχία της Τινησίας εξαρτάται από την οικονομική της επιτυχία. Αυτά, τα δυο πάνε παρέα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το υποστηρίσουμε και η υποστήριξη των επενδύσεων παίζει σημαντικό ρόλο. Οι διαπραγματεύσεις για μια βα... Ε, βαθιά... βαθύτερη συμφωνία ε, ελευθέρων συναλλαγών και εμπορίου ε, συμβαδίζει με την οικονομική ανάκαμψη της Τινησίας αλλά και με την μεταρρυθμιστική πορεία στην οποία έχει μπει η Τινησία και πρόσφατα πήγα στην Τινησία το περιορισμένο φθινόπωρο για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσει για την βαθύτερη αυτή συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι δεδομένη τη ευάλωτη οικονομική κατάσταση, οι διαπραγματεύσει αυτέ είναι τεράστια πρόκληση για την Τινησία. Γι' αυτό προτείνουμε, όπω είπε και η συγγήτρια, μια ασυμμετρική και σταδιακή προσέγγιση στο άνοιγμα τη αγορά σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Στι ε, Τινησιακέ Αρχέ είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε σε στάδια. Μια καλή διαπραγμάτευση ξεκινά από την αμοιβαία συνεννόηση όπου πρέπει να ενσωματωθούν οι πραγματικότητες, οι διτηρότητες και οι προσδοκίες αλλήλων. Ε, έτσι θα πρέπει να ε, φτιάξουμε ένα πακέτο το οποίο θα στηρίξει την μεταρρυθμιστική πορεία και θα αναβαθμίσει ορισμένους τομείς κλειδιά όπως η γεωργία και οι υπηρεσίες αλλά θα παρέχει και στήριξη στον ιδιωτικό τομέα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη σημασία της ε, νησιακής κοινωνίας των πολιτών. Έχουν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην μεταρρυθμιστική πορεία της ε, νησίας. Θα πρέπει επίσης να παίξουν ρόλο και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, πολλές επαφές είχα όταν ήμουν στην νησία και είχαμε διάλογο για την βαθύτερη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Είμαι ευτυχής που υπάρχει διαφάνεια και διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, των, της νησίας αλλά και των ευρωπαϊκών οργανώσεων όπου η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων. Η στενή και η διαρκή συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών θα παίξει ρόλο για να υπάρξει γνώση για τι διαπραγματεύσει και για τη μελλοντική εφαρμογή του. Όσον αφορά τώρα το ελαιόλαδο, στόχο του μέτρου είναι να στείλουμε θετικά πολιτικό μήνυμα προ την Τινησία και να ε, επιφέρουμε ένα απτό συγκεκριμένο όφελο στην οικονομία ε, που δημιουργώντα και θέσει απασχόληση που είναι τόσο απαραίτητε και καλωσορίζω την εργασία για την, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επενώ την εργασία της εισηγήτριας κυρία Τεσσαρνές και όλων των ε, συνεισηγητών, σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω πως αύριο θα υποστηριχθεί η πρόταση αυτή από την Επιτροπή Ίντα ώστε το όφελος που προσφέρουμε στην την να μπορέσει να αρχίσει να ε, ισχύει χωρί περαιτέρω καθυστέρηση. Οι εισαγωγέ ε, λεολάδου βεβαίω θα πρέπει να συμβαδίζουν με την προτιμησιακή προέλευση και με τι υγειονομικέ και φυτογειονομικέ απαιτήσει. Το μέτρο προτείνεται για μια περιορισμένη χρονική περίοδο, μια διετία και θα παρακολουθείτε στενά. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το σύνολο της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ελαιολάδου. Αυτός ο όγκος ποσόστασης θα απορροφηθεί σύμφωνα με την κατάσταση της αγοράς χωρίς σημαντικό αντίκτυπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την εργασία που έχουμε κάνει, που έχετε κάνει σε αυτό το θέμα και ελπίζω πως αύριο θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε στο πλευρό του την Ισιακού Λαού, είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε βράχει μέσω και μακροπρόθεσμα, μέσω της ε, εταιρική σχέσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Tak, ε, dziękuję. Ε, a teraz w imieniu Komisji Rolnictwa. κυρία Καρσία. Κιλέρα Καρσία, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μάλστρομ, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Ντεσσαρνές για την έκθεσή της, αλλά εγώ ήμουν εισηγήτρια για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και θέλω να την διαβιβάσω εδώ, γιατί νομίζω ότι δεν την έχετε λάβει αρκετά υπόψη, ούτε έχει αναγνωριστεί. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η Επιτροπή Γεωργίας ε, ήταν υπέρ αυτής της πολιτικής συμφωνίας για τα έκτακτα μέτρα, τα εμπορικά με την Τινησία. Σαφέστατα έγινε μια ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία ήταν υπέρ ε, της απόρριψης, της πρότασης. Λοιπόν, η, Γεωργία, η Επιτροπή Γεωργίας είναι υπέρ της πολιτικής συμφωνίας, αλλά ειλικρινά σας λέγω ότι δεν διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των παραγωγών στην Ευρώπη με τρόπο σωστό. Πολλέ ζώνε τη υπαίθρου και η περιοχή μου η Ανδαλουσία εξαρτώνται πάρα πολύ από την παραγωγή του λαδιού. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ελαιόλαδο. Και παρακαλώ την Ολομέλεια και τους παρόντες και σας κυρία Επίτροπε να δείξετε ευαισθησία και να βάλετε τις τροπολογίες 11, 12, 13 και 14 και τελειώνω, Πρόεδρε. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι τροπολογίες αυτές δεν βλάπτουν καθόλου τη συμφωνία ούτε την υποστήριξή μας για την Τινησία που είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων ακολουθούν τώρα. Εξ ονόματο του ΕΛΚ, πρώτος ο κύριος Σαντιάγκο Φίσας. Εξέλα. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε η Τινησία είναι η μόνη μάλλον χώρα της ε, Μεσογειακής Λεκάνης που βρίσκεται στον δρόμο μιας πραγματικής δημοκρατίας. Αυτό που είναι καλό παράδειγμα για όλο τον αραβικό κόσμο είναι κακό παράδειγμα για τους ε, ε, φανατικούς Ισλαμιστούς που κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστραφεί η χώρα και να αποσταθεροποιηθεί. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στην δυνησία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και στηρίζω καθολικά αυτή την πρόταση για αύξηση των ποσοστώσεων εισαγωγή αδασμολόγητου ελαιόλαδου από την Ισία. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτούμε τι συνέπειε. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ισορροπίες, υιοθετώντα μέτρα που θα εγγυηθούν ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί ελαιόλαδου δεν θα βγουν ζημιωμένοι από αυτή τη συμφωνία. Ω προ αυτό, Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες που διευκρινίζουν αυτό το σημείο και που ελπίζω αύριο θα υπερψηφιστούν. Όπως λέει και το κείμενο που αύριο θα ψηφίσουμε, αυτή η παραχώρηση εκτάκτων μέτρων δεν καθορίζει την πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία, που την οποία στηρίζω απόλυτα και θεωρώ πως είναι ακόμα ένα βήμα στην δρέωση της δημοκρατίας στην Ισία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών, ο κύριος Εμμανουέλ Μορέλ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω πως ε, σε όλα τα έδρανα αυτού του σώματος έχουμε ε, έναν ίδιο στόχο, ε, δηλαδή να βοηθήσουμε συγκεκριμένα και ε, με διάρκεια, σε διάρκεια την Τινησία και τον Αρδενισιακό λαό. Υπόθηκε, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε και να το θυμίσουμε γιατί είναι σημαντικό για εμάς τους Ευρωπαίους. Είναι η Τινησία, το Λίκνο και το σύμβολο της Αραβικής Άνοιξης. Είναι από τις λίγες χώρες σήμερα που πετυχαίνει την μετα... δημοκρατική μετάβαση. Αλλά βεβαίως και η κυρία Ντεσανέ σωστά το θύμισε, έχει να αντιμετωπίσει τεράστια πολιτικά, πολιτικές προκλήσεις με την τρομοκρατική περιβαλλοντική απειλή, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις με μαζική ανεργία, τον τουρισμό που καταραίει. Εν ολίγης, ε, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα και με διάρκεια τους ταινίσιους. Οικονομικές έκτακτες βοήθειες. Ε, πολλά κράτη-μέλη δεσμεύθηκαν γι' αυτό. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα, επιγόντως και προσωρινώς, είναι η ε, επέκταση των ποσοστώσεων εισαγωγής αδασμολόγητου ελαιόλαδου. Και εδώ δεν πιστεύω, δεδομένης της μικρής σημασίας του την Ισιακού Ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Αγορά ότι θα επηρεάσει τις τιμές του τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Είναι ένα προσωρινό επίγον μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει λίγη ανάσα στην, Ευρω... στην Ισιακή οικονομία. Και έπειτα υπάρχει και αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Καταρχήν πρόκειται για μια εταιρική σχέση. Εταιρική σχέση που δεν είναι μόνο οικονομική φύση αλλά και πολιτική φύση. Και αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι συμμετρική, δεν είναι σταδιακή η συμφωνία αυτή, αλλά και εδώ θα πρέπει, και εδώ απευθύνομαι στην Επίτροπο που το γνωρίζει, γνωρίζει νομίζω ότι θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να δείχνουμε εκτίμηση στην κοινωνία των πολιτών που κάποιες φορές έχει δίκιο να ανησυχεί και πρέπει να την καθησυχάσουμε και να πούμε ότι η Ευρώπη σε αυτή τη συμφωνία αποδεικνύει ότι δεν συνηθίζει τη δουλειά της σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά ότι γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να τη λάβει υπόψη. Πρέπει να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά και στο ύψος των προσδοκιών του λαού της Τινησίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ECR, ο κύριος Νότης Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ενώ η Τρόικα φτωχοποιεί τους Έλληνες αγρότες και διαλύει τον αγροτικό τομέα, ενώ οι δανειστές επιβάλλουν σκληρή φορομπηκτική πολιτική κατά του αγροτικού κόσμου και διαλύουν το ασφαλιστικό του σύστημα και τον ΟΓΑ, ενώ οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από τα έντονα περσινά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την παραγωγή τους, την ίδια στιγμή έρχεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί αδασμολόγητη ποσόστοση εισαγωγής 70.000 τόνων τυνησιακού λαδιού για το 2016 και 2017. Η ενέργεια αυτή της Ένωσης αποτελεί ταφόπλακα για τους στοχοποιημένους Έλληνες παραγωγούς που ήδη βλέπουν τις φετινές τιμές του λαδιού τους να καταραίουν. Γιατί άραγε η νομοθετική πρόταση εφαρμόζει την αδασμολόγητη εισαγωγή τυνησιακού λαδιού αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ποιους θέλει να καλύψει, Ποιους θέλει άραγε να ευνοήσει, κυρία Μάλστρομ, η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης, η ελαιοπαραγωγή της Λέσβου, του νησιού που κατακλείζεται από χιλιάδες πρόσφυγες, δεν αντέχουν άλλο χτύπημα κάτω από τη μέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, on behalf ALDE. ALDE τώρα. κυρία Για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο και του συναδέλφου. Υποστηρίζουμε τη στενατρή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία μέσω του εμπορίου, αναγνωρίζοντα ε, ε, τα θέματα που αντιμετωπίζει ο λαό στην την Ισία. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλε οι προκλήσει σήμερα και μα ενθαρρύνουν οι συνεχιζόμενοι αγώνε να καταπολεμήσουν την ε, καταπίεση, την αυταρχική ή την ισλαμική και τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Τινεσία είναι και θα πρέπει να είναι ένα υπόδειγμα για αυτή την ειρηνική μετάβαση. Ωστόσο, είναι δύσκολος ο δρόμος προς την Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ο πρώτος και ουσιαστικός εταίρος της ε, Τινησίας. Και να θυμηθούμε γιατί πριν από πέντε χρόνια ο Μουχάμεντ Βαζίζη σε μία ε, δράση, σε μία ε, δράση που φανέρωνε την απελπισία του, αυτό και έγινε ένα σύμβολο κατά της ε, διαφθοράς και της καταπίεσης οποιασδήποτε ευκαιρίας για τους νέους ιδιαίτερος. Και πιστεύω ότι μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία θα συμβάλλει στην εξέλιξη, ανάπτυξη και ελευθερία της Τινησίας για να μπορέσει ο λαός να διαμορφώσει το μέλλον του. Και καλό τους ε, συναδέλφους να μην ε, αντισταθούν και να μην καταψηφίσουν μια ελάχιστη ποσόστοση σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο. Θα είναι ελάχιστη. Ελάχιστο ο αντίκτυπο στην Ευρώπη, ενώ θα είναι πολύ μεγάλο και θετικό στην Τινησία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα από την QNGL, ο κύριος Λεγερίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το είπε και η κυρία Ντεσανέζ. Η ευθύνη μας είναι να είμαστε συμπαραστάτες στο πλευρό της δίκης χειραφέτησης του τυνησιακού λαού που γίνεται, ε, το είπαν πολύ ε, με μεγάλες δίνες και ε, δεινά από την τρομοκρατία που χτύπησε τη χώρα τρεις φορές με τεράστιες ολέθριες συνέπειες. Προτιμησιακές σχέσεις μπορούμε να αποφασίσουμε λαμβάνοντας υπόψη τους ευαίσθητους τομείς έρθον της Μεσογείου. Ε, φρούτα και λαχανικά ε, όπου θα πρέπει να έχουμε χρονοδιαγράμματα παραγωγής για να μην έχουμε καταστροφικό ανταγωνισμό και το ίδιο ισχύει για την προστασία της παραγωγής ελαιολάδου. Ε, όταν έχουμε πλήρης ελεύθερες συναλλαγές ε, που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς διαφωνούμε, προσπαθούμε και προτιμούμε να έχουμε πραγματική συνεργασία που θα αποφασίσουμε μετά από διαβουλεύσεις με την κοινωνία της Τινησίας και μελέτες αντικτύπου για να προετοιμαστούν αυτές οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά. Εξ ονόματος των Πρασίνων το λόγο έχει ο κύριος Γιώργη Σεμπαστιά. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πίτροπε. Και πάλι συζητούμε εδώ για τη δυνησία και τώρα για πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Φαίνεται ότι αρχίζει να σχηματίζεται αυτή η δυνατότητα, η εικόνα, ότι είναι ο μόνος δημοκρατικός εταίρος μας στη Βόρεια Αφρική και θα πρέπει χωρίς όρους να υποστηρίζουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μια έχουμε έκτακτα εμπορικά μέτρα για να μπορούμε να εισάγουμε περισσότερο ελαιόλαδο αδασμολόγητο. Είμαστε απολύτως υπέρ και σας το λέω εγώ που είμαι από μια χώρα που παράγει πάρα πολύ λάδι και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Γιατί θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να βοηθούμε την νησία που τόσα υποφέρει στον δρόμο για τη δημοκρατία. Η τρομοκρατία, η κρίση με τους ε, μετανάστες που έχει από τη Λιβύη κτλ. Ε, αντί να βοηθήσουμε συγκεκριμένα, γιατί δεν έχουμε μεγάλη φαντασία, μιλάμε και πάλι για Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, με μεγάλες ανισορροπίες. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι μικρή η οικονομία με διαρθρωτικές ελλείψεις και αδυναμίες ή την Ισία. Να έρθουν οι τινήσει στην Ευρώπη, λέμε, αλλά έρχονται μόνο όταν έχουν βίζα. Εμεί χωρί θεωρήσει μπορούμε να πάμε στην Ισία δεν υποστηρίζει η κοινωνία της Τινησίας τέτοιου είδους συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσουμε τους γειτονές μας. Εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε τα δόγματά μας του νέου φιλελευθερισμού και να επιβάλλουμε μια οικονομία σε μια χώρα που δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Η πολιτική και η οικονομική στήριξη γιατί θα πρέπει να είναι τόσο ανισόρροπες. Ευχαριστώ πολύ. Eh, e Σας ευχαριστώ από το EFD τώρα. Ο κύριος Δαμάτο. Η, κυρία Δαμάτο. Για ένα μισό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ας μην κάνουμε αυτό το τεράστιο λάθος. Δεν θα βοηθήσουμε το λαό της Τινησίας με μηδενικές, ε, μηδενικούς δασμούς για το Ελλάδα. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να καταστρέψουμε την γεωργία στο νότο της ε, Ευρώπης. Μην το κάνουμε λοιπόν αυτό στους καταναλωτές μας και στους παραγωγούς μας. Ακούστε τα λόγια τη Επιτροπή Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσοχή. Υπάρχει κίνδυνο ε, παραποίηση του Made in Italy και απάτη ει βάρο των καταναλωτών. Στον Ιταλικό γεωργικό τομέα επιβάλλεται μια ανιωστή ε, απόφαση χωρί να λαμβάνεται υπόψη αντίκτυπο σε οικονομικό, εργασιακό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι από τη στιγμή που θα έρθει στο ευρωπαϊκό λιμάνια κάποιο πονηρό θα μετατρέψει σε Ιταλικό λάδι το νησιακό ε, δεν είναι εύκολη η ανείχνευση και αυτό το λέω μετά από ε, την κατάσχεση 5.000 ε, τόνων στην Απουλία ε, χρησιμοποιείται από κάποια εταιρεία που ε, κερδίζει ανακατεύοντας τα λάδια. Η γεωργία της Νότιας Ευρώπης φέρει το βάρος του εκδημοκρατισμού των χωρών της Βόρειας Αφρικής, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ισία να αγωνιστεί κατά της φτώχειας και του Ισλαμικού φονταμενταλισμού βεβαίως, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ευρωμεσογειακή γεωργία που να αξιοποιεί την δική μας γεωργία και όχι μόνο να στηρίζει ε, που και που. Κύριοι Ιταλοί Ευρωβουλευτές, ε, με την θετική σας ε, ψήφο στην εισαγωγή την Ισιακούλα Διού, εσείς βάζετε φωτιά σε έναν πόλεμο ανάμεσα στους στοχούς. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Κάσπαρη. Μπλε κάρτα από τον κύριο Κάσπαρη, τη δέχεστε. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, κύριο Κάσπαρη. Uh, Αξιότιμοι συνάδελφε, μιλήσατε για τις αρνητικές επιπτώσεις ενδεχομένως ε, στην ηλεκτρομηχανία στην ε, Ιταλία. Συμφωνείτε ότι η αγορά ε, στην Ευρώπη ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια τόνους και μιλάμε για 35 εκατομμύρια τόνους επιπλέον από την Φινησία. 5.000 τόνους από την ε, την Ισία. Αν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε την ε, γεωργία στην την Ισία, να φροντίσουμε να ε, εισαγάγουμε λίγο το ελαιόλαδο και να μην εμποδίζουμε αυτό το μικρό ποσοστό, το μικρό κλάσμα που εισαγάγεται από την Τινησία. Αυτό που είπα εγώ είναι τελείως διαφορετικό. Μίλησα για ευρωμεσογειακή γεωργική πολιτική. Αυτό σημαίνει η συμπερίληψη και των χωρών της Βόρειας Αφρικής. Σημαίνει ότι όλη η παραγωγή, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε, δεν, τα προϊόντα είναι τα ίδια. Γι' αυτό ε, μιλώ για πόλεμο ανάμεσα στους στοχούς θα πρέπει να θυμίσουμε ότι πέρα από τους 35.000 τόνους επειδή έχουμε άλλους 56.000 τόνους που στην ουσία έχουν πάρει χάρη, ας το πούμε έτσι, είναι αδασμολόγητα δηλαδή, ε, αδασμολόγητες εισαγωγές. Ε, δεν λέω να μην τους βοηθήσουμε, όχι. Είπαμε ότι ένα οχυρό της, ε, της δημοκρατίας θα πρέπει να το βοηθήσουμε όπως η Τινησία, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταμάτο. Ο κύριος Λουαζό. Oui, ναι, κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο σχόλια να πω για την πρόταση αυτή. Πρώτον, για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό το μανδύα της υποστήριξης του εκδημοκρατισμού ανακατεύεται σε μια χώρα που τη χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά. Είδαμε τι έγινε και πώς αναμίχθηκαν κάποιες χώρες στον εκδημοκρατισμό των χωρών της Βόρειο Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής. Με αντίκτυπο, ε, τι, θα βοηθήσει το ελαιόλαδο τώρα για την πολιτική κρίση. Ενώ θα πλέξει τους Ευρωπαίους ελαιοπαραγωγούς. Γνώρισαν μεγάλες κρίσεις και δεν το έχουν ανάγκη τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδεινώσει την κατάσταση για πολιτικούς λόγους. δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και άλλα δεινά. Όπως συχνά το Κοινοβούλιο ε, οργανώνει τον αθέμητο ανταγωνισμό γιατί είναι αδεσμολόγητες οι ποσότητες αυτές και οι μικροκαλλιεργητές και πάλι θα είναι τα κορόιδα της υπόθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει θέλει να δείξει ελεγγύη εις βάρος των καλλιεργητών της Νότιας Ευρώπης. Η κοινή λογική επιβάλλει να εγκαταλειφθεί η πρόταση γιατί θα είναι βάρος ε, του ευρωπαϊκού γεωργικού κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Τσίκου για μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να πω με σαφήνεια ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ μιας πολιτικής ε, που υποστηρίζει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Τινησίας και στηρίζει το Τινησιακό σύστημα. Αντίθετα, είμαι κάθετα αντίθετος από την υιοθέτηση τέτοιου είδους διατάξεων σε σχέση με τον ε, ε, ελαιόλαδο. Όχι όμως για το ελαιόλαδο συγκεκριμένα. Είμαι κατά μιας πολιτικής που τη μια διαλέγει το ελαιόλαδο, την άλλη την ντομάτα, την άλλη το κρασί, την άλλη όλα όσα παράγονται μόνο σε ορισμένες περιοχές. Γιατί να μην μιλήσουμε για το γάλα, γιατί να μην αρχίσουμε να μιλάμε για το κρέας, γιατί δηλαδή να μην γίνεται η διαφοροποίηση αυτού του βάρους που μόνο τη δικά μας νότιες περιοχές, Σικελία, η Απολία, η Σαρδινία ε, παράγουν. Καταστάσεις όπως σήμερα έχουν γονατίσει. Γιατί εδώ δεν θέλουμε ε, να δούμε πόσο παράγουμε. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε ποια ζημιά ε, θα επιβαρύνει τους μικρούς παραγωγούς μέσω τέτοιου είδους πολιτικών. Και προσθέτω ότι η αξιοπιστία της Ευρώπης χάνει και, γίνεται ακόμα, και πλήττεται ακόμα περισσότερο από τη δυνατότητα να δώσει ένα, από την αδυναμία μάλλον να δώσει ένα έντονο μήνυμα συνοχής ακριβώς λόγω τέτοιου είδους ε, ε, ε, μέτρων. Και γι' αυτό έχω προτείνει και σχετική τροπολογία για απόρριψη της πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίκτορ Μποστινάρο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρία εισηγητρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγητρία για την εξαιρετική της έκθεση και Σύμφωνο και την υποστηρίζω απόλυτα. Η Τινησία είναι μια πηγή ελπίδας για όλους μας. Αλλά η Τινησία σήμερα βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων οικονομικών, κοινωνικών και προκλήσεων ως προς την ασφάλεια της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κατεπηγόντως να δράσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη. Τώρα χρειάζεται υποστήριξη και αλληλεγγύη, όπω άλλωστε υποσχεθήκαμε στο παρελθόν και την υπόσχεση αυτή δεν την έχουμε τηρήσει επαρκώ. Τα αυτόνομα αυτά εμπορικά μέτρα για την, την συγκαταλέγονται σε αυτό το πακέτο των κατεπηγόντων μέτρων που έχουμε υποσχεθεί στην Τινησία. σας. Σα παρακαλώ λοιπόν υποστηρίξτε το κείμενο όπω προτείνεται από την εισηγήτρια. Να αποφύγουμε να προκληθεί ζημία στην ε, την Ισία λόγω μεμονωμένων συμφερόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το ελαιόλαδο αποτελεί ένα σημαντικό αγαθό εξαγωγής για την Ισία. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντική η διάταξη αυτή για την χώρα. Σελιμοβίτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τινησία είχαν ε, τεράστιο αντίκτυπο στην Τινησία και στην ήδη ασθενή οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν και η πρότασή της για επιπλέον εξαγωγές ελαιόλαδου είναι κάτι που καλωσορίζουμε. Κάποιοι παραπονιούνται για τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν αυτές οι επιπρόσθετες εξαγωγές. Αλλά οι ρυθμοί μιλούν από μόνοι τους. Αυτό το ποσό το, το καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι κάθε χρόνο. Έχουμε αύξηση κατά 50% την παραγωγή και το ποσό που θα μάλλον ο όγκο ελαιόλαδου που θα λυθεί από την τελικά θα είναι 1,7%. Ερωτώ λοιπόν αυτού του βουλευτέ, αυτό το 1% επιπλέον, πώ θα καταστρέψει αυτή την ευρωπαϊκή την αγορά που υπάρχει έλλειψη 48% αλλά να σας πω ότι στην Τινησία ένα εκατομμύριο άνθρωποι απασχολούνται στην παραγωγή ελαιόλαδου, μεγάλο και το βασικό ε, αγαθό εξαγωγών της Τινησίας. Για μας δεν είναι τίποτα, γιατί την Τινησία είναι πάρα πολύ μεγάλο όμως το θέμα και ελπίζω το Κοινοβούλιο να επιδείξει την αλληλεγγύη που είχε υποσχεθεί αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Φορέντσα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με το στόχο που λέει ότι θέλει να επιδιώξει η Κομισιόν να βοηθήσει την δημοκρατία της Τινησίας και την οικονομία της που έχουν πληγεί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. επίση είμαι υπέρ οποιασδήποτε πρακτικής οικονομικής και πολιτικής αλληλεγγύης με τους λαούς της Μεσογειακής Λεκάνης. Ταυτόχρονα όμως ε, πολύ με δυσαρεστεί αυτό το μέσο που προτείνεται. Συμφωνία ελεύθερων συλλαγών και μηδέν δασμοί για την εισαγωγή του ελαιόλαδου. Η απελευθέρωση δεν είναι το μέσο για να αναπτυχθεί η ε, αναπτυσσόμενη οικονομία. Μάλιστα θα μπορούσε να βοηθήσει τον ε, λαό της νησίας η ακύρωση του χρέους, η διαγραφή του χρέους. Νομίζω πως είναι, ε, γίνεται μια ρητορική προσπάθεια για βοήθεια των παραγωγών της Ισίας ενώ έτσι βοηθούνται μόνο οι μεγάλες εταιρείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελαιόλαδο κυρίως το νότιο, όπως, στην Νότια Ευρώπη όπως στην Απουλία, παραγωγή εκεί έχουν ε, πληγεί από τα βακτήρια αλλά και από την ε, συμφωνία για την εισαγωγή του ελαιόλαδου. Εγώ θα καταψηφίσω όχι μόνο για να βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι και οι, οι παραγωγοί αλλά και οι τινήσιοι. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κασπάρη. Για ένα λεπτό. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Τινησία, αλλά περιμένουμε και κάτι α, να μας δώσει την Ισία. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Τινησία. Με επιπρόσθετες ε, ποσοστώσεις για ελαιόλαδο. Χαμηλές σε σχέση με την ε, ευρωπαϊκή παραγωγή και θέλουμε να δώσουμε μια σωστή και καλή ε, συμφωνία εμπορική για να δώσουμε μια προοπτική στην Τινησία. Αλλά πρέπει και την Τινησία να πάρει στα σοβαρά τι υποχρεώσεις τη. Και βλέπω στην παρούσα φάση ότι πολλοί Τινήσοι φεύγουν και έρχονται γιατί στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι ε, με δυσκολία αποδέχεται ε, την επιστροφή πρόσφυγες στην Τινησία που δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εδώ. Στο 2015, για παράδειγμα, στη χώρα μου δεν υπήρχε ούτε ένα ενίσιος μετανάστευση του, ο οποίο να αναγνωρίθηκε ως πρόσφυγα. 0,0%. Όταν, ε, αν λοιπόν αγγιηθούμε αυτέ τι εμπορικέ ποσοστώσεις, ελπίζω η Τινησία να δείξει μεγαλύτερο πνεύμα συνεργασία και να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσπαρη. τώρα το λόγο έχει η κυρία Αρένα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, κυρία Συγγήτρια. Είναι γεγονός ότι αυτή η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σε μια περίεργη κατάσταση από την επανάσταση του 2011, αλλά και πριν θα έλεγα, η Τινησία χρειάζεται βοήθεια. Και χαίρομαι για τη συμφωνία για το ελαιόδαδο. Καμιά φορά εκπλήσωμαι από την αμυντική γραμμή κάποιων συναδέλφων εδώ. Ε, που ταράζονται για το 2% και λιγότερο ε, της παραγωγής ελαιολάδου στην Ευρώπη, ενώ καμιά φορά όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που θα μπορούσαν να έχουν πολύ πιο ελεύθερες συνέπειες στη Γεωργία, είναι οι μεγαλύτεροι και οι πιο ένθερμοι υπερασπιστές τους. Λοιπόν, για να ξαναδούμε τι θα χάσει ενδεχομένω η Γεωργία. Ε, στη συμφωνία αυτή θα πρέπει να προσέξουμε το εξή θα έλεγα εγώ. Θα πρέπει να δημιουργούνται ε, ποιοτικέ δουλειέ για η φόρο ανάπτυξη στην Τινησία. Θέλει προσοχή, γιατί η συμφωνία αυτή λαμβάνει υπόψη την ε, διαφορεία που υπάρχει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και το είπατε εσείς ε, κυρία Επίτροπε να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών γιατί έχει πολλές προφορίες να μας δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βουλευτά ο κύριος Σαλβατόρε Ντομένικο Πουλιέζε. Πολιέζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως δεν μπορεί κανείς ένα μεταξύ μας να μην είναι αλληλέγγυος με τον λαό της Τινησίας μετά από τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της περισμένης χρονιάς. Όμως η Ευρώπη μετατρέπει το δικό της ε, μέρος μέσω της ε, χορήγησης 500 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση για να στηριχθεί η νεαρή ε, δημοκρατία της Τινησίας αυτά τα 70.000 τόνους ελαιόλαδου που προστίθεται, όπως κάποιος θύμισε, στις 56.700 τόνους που ήδη προβλέπονται από την ισχύουσα συμφωνία, δεν γίνεται άλλο παρά να σφαγιαστεί η γεωργία της Νότιας Ευρώπης και κυρίως της Ιταλίας, με ιδιαίτερο τρόπο και σε μια φάση που η ασθένεια, η ξυλέλα που ε, έπληξε τα ρίζες της Ιταλίας μείωσε κατά 47% το σύνολο της παραγωγής της Ιταλίας. Γι' αυτό και δεν θα υπερψηφίζω αυτή τη διάταξη για να μην συνεχίζεται Γι αυτό η σφαγή της γεωργίας της Νότιας Ευρώπης. Ευχαριστώ. Παντσέρι ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την κυρία Ντισαρνές για την εργασία της, ε, για την κατάσταση στην Ισία ήδη πιώθηκαν πολλά. Εγώ πιστεύω πως ε, καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει σημαντικά πολιτικά, οικονομικά για να μπορέσει αυτή η μετάβαση να ολοκληρωθεί θετικά και θα πρέπει αυτό να γίνει σε το χρόνο. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο. Τώρα οι διαπραγματεύσει για, ε, για την εμπορική συμφωνία θα πρέπει αυτή την κατεύθυνση να ακολουθήσουν ώστε να υπάρξει ε, θετικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία τη Τινησία. Η συμφωνία θα πρέπει να βασιστεί στη μέγιστη διαφάνεια και να εμπλέξει στον μέγιστο βαθμό την κοινωνία των πολιτών τη ε, Τινησία. Αυτό το ζητάμε εντόνω και αποφασιστικά. Σε αυτό θα πρέπει να μπει και η απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εισαγωγή των επιπλέον ποσοστώσεων. Τέλος, πιστεύω πως μπορώ να πω πως η Τινησία περιμένει από το Ευρωκοινοβούλιο ένα μήνυμα σημαντικό για να ορίσει ένα πλαίσιο ε, ισορροπημένων εμπορικών σχέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρούας, για δύο λεπτά. Για ένα λεπτό, ευχαριστώ. Φυσικά είμαστε υπέρα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες ε, και ιδιαίτερα στην, ε, για την Τινησία. Ωστόσο, θα είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά την μορφή αυτής της αλληλεγγύης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι μόνο γιατί ακόμη μια φορά πλήττεται ένας τομέας ε, της ε, ευρωπαϊκής παραγωγής αλλά ε, γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνονται άλλες προσπάθειες μέσω των υπολείπων πολιτικών γυτνίασης, συνεργασίας κτλ. Παράλληλα, γνωρίζουμε πόσο πλήττονται οι οικονομίες των μεσογειακών χωρών της Ένωσης όπως της Πορτογαλίας. Γι' αυτό το λόγο η αρχή της αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για ε, τις χώρες εκτός της Ένωσης αλλά και για μέσα στην Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε τις οικονομίες των κρατών μελών και να ψάχνουμε εναλλακτικέ δίκες για να στηρίξουμε τις οικονομίες των τρίτων χωρών στην ε, ψηφοφορία. Ε, θα σκεφτώ ποια θα είναι η θέση μου για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ κύριο Σπαρνιό. Ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Μεγάλη πρόκληση ε, στην ευρωπαϊκή γειτονία, το καταλάβαμε όλοι, η, την Ισία. Πώς θα τη βοηθήσουμε. Η πρώτη δράση που απαιτείται είναι να αυξηθούν οι εξαγωγές της προς εμάς, ιδιαίτερα στον ε, κομβικό αυτό τομέα του ελαιολάδου. Μα είναι προφανές αυτό. Και μετά θα πρέπει γρήγορα να συνάψουμε εταιρική σχέση για δίκαιες συναλλαγές Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ισίας. Θα πρέπει όμως η στήριξή μας να πάει παραπέρα και το θέμα της ασφαλείας αξίζει ευρεία περιφερειακή συνεργασία με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό και ειδού ένα πεδίο δόξης λαμπρό για να επενδύσει όλη τη διπλωματική ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, η στήριξη της οικονομίας είναι η στήριξη της δημοκρατίας στην κατά πολέμηση της δημοκρατίας που την πλήττει. πολέμηση της δημοκρατίας σημαίνει ότι θα προστατεύουμε τους αυτούς μας. Ιδού το μήνυμα θα πρέπει όλοι απόψε να ακούσουν εδώ μέσα σε αυτό το εμικύκλιο. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Λαβία. Grazie, Ευχαριστώ. Εγώ θα καταψηφίσω την πρόταση. Διότι οι στόχοι της πρότασης είναι σωστοί, αλλά τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιτευχή των ίδιων στόχων είναι λάθος. Η μείωση των δασμών στις εισαγωγές δεν φέρει κανένα όφελος στους τινήσιους παραγωγούς και ούτε στους οικονομικούς παράγοντες της χώρας. Θα ωφελήσει μόνο μια ομάδα ε, Ευρωπαίων εισαγωγέων ελαιολάδου που θα πλουτίσουν με τους φόρους που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι αυτή η σωστή πολιτική, ούτε είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Νομίζω μάλιστα πως ακολουθούμε λάθος κατεύθυνση. Όχι μόνο τιμωρούμε ακόμη μια φορά τον γεωργικό τομέα της Νότιας Ευρώπης και μάλιστα με σοβαρό τρόπο, αλλά κάνουμε μια δράση που δεν θα έχει κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το καλό λάδι είναι διάφανο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα πολύ πολύ θολό λάδι. κύριος Δικάστρο. Δεκάστρο, με συγχωρείτε. Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, το να βοηθηθεί η Τινησία σε αυτή την τόσο δύσκολη φάση είναι ηθικό καθήκον και δεν θέλουμε βεβαίω να κάνουμε πίσω. Ωστόσο, πιστεύουμε πω θα υπήρχαν άλλοι τρόποι πιο συγκεκριμένοι και αποτελεσματικοί να βοηθηθεί η οικονομία τη Γεωργία τη Τινησία. Α πούμε, μέσω προγραμμάτων αξιοποίηση του Τινησιακού ελαιολάδου, που είναι εξαιρετικό προϊόν και που ήδη εισάγεται σε μεγάλε ποσότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, οι ίση εξέφρασαν αμφιβολίες γιατί αυτά τα μέτρα θα εφαλίσουν τους Ευρωπαίους εμπόρους και πολύ λίγο τους Τινήσιους. Ε, αυτά όλα δεν είναι αποτέλεσμα ε, κάποιες κορπορατίστικης ε, στάσης. Όχι. Είμαστε, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι αυτού του μέτρου και ποιοι θα ωφεληθούν. Θα θέλαμε διαφορετική συμπεριφορά. Τουλάχιστον όμως συζητώ από τους συναδέλφους να στηρίξουν τις τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας που αμβλύνουν κάπως τις πτώσεις τρέβλωσης στην ευρωπαϊκή αγορά αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πιτήρη, Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Τινησία είναι μία από τις σπάνιες εκείνες χώρες όπου μετά την ε, ε, Αραβική Άνοιξη δεν προκληθήκε χάος όχι. Ανταυτού αυτό υπήρξε μια δημοκρατική μετάβαση. Θα πρέπει λοιπόν για το λόγο αυτό να βοηθήσουμε την, την Ισία να διατηρήσει αυτή την ευάλωτη και ευαίσθητη δημοκρατία που έχει πετύχει και να ε, προωθήσουμε τα Ισιακά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά όχι με μέτρα τα οποία θα βλάψουν την αγορά της Ευρώπης, όπως έγινε με το ρωσικό εμπάρκο, για παράδειγμα. Το ελαιόλαδο είναι το πιο σημαντικό αγροτικό προϊόν που εξαγαγεί την Ισία και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται υποστήριξη αυτή. Αλλά η εισαγωγή ελαιόλαδου από την Τινησία θα δυσκολέψει την κατάσταση και τη ρύθμιση της αγοράς ελαιόλαδου στην Ευρώπη. Γιατί θα διαπιστώσουμε ότι θα υπάρξει και επιδείνωση της ποιότητας ελαιόλαδου και εκτός αυτού έχουμε αρκετό ελαιόλαδο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την, ε, την Ισία, αλλά για το συμφέρον των ε, Κροατών και των Ευρωπαίων παραγωγών θα πρέπει να είναι περιορισμένη αυτή η υποστήριξη. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, α αρχίσουμε από το πιο σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είχε την πολιτική υποχρέωση να είναι πιστή στην ε, υποχρέωσή τη να ενισχύσει τις εμπορικές σχέση με την Τινήσια Τώρα έχει και την ηθική υποχρέωση να στηρίξει ακόμη περισσότερο την Τινησία μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν πολύ σοβαρά την οικονομία της χώρας. Γι' αυτό έχει νόημα το να στηριχθεί ο τομέας του ελαιολάδου της Τινησίας. Αν και πρέπει να λάβουμε επίση υπόψη ότι το τομέα του ελαιόλαδου είναι ένα τομέα σημαντικό για πολλέ χώρε τη Νότια Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σαφή τα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, τα μέτρα αυτά είναι εξαιρετικά, προσωρινά, ε, δεν θα διαρκέσουν πάνω από δύο χρόνια. Δεύτερον, όπως προτείνει η συγκεντριά μας, θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα αξιολόγησης ε, που θα επιτρέπουν την ε, αναστολή του σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρή διαταραχή της ευρωπαϊκής αγοράς ελαιολάδου. Να έτσι θα είμαστε αλληλέγγυοι με την Ισία όπως είναι το καθήκον μας, αλλά θα έχουμε και την απαραίτητη ηρεμία στον ευρωπαϊκό τομέα ελαιολάδου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται ο κατάλογος των και τώρα περνάμε στη δικασία Catch Σε έναν Σεράνο ε, η Τινησία περνά μια περίοδο μεγάλων ανταδροχών και αξίζει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το επιπλέον ποσόστοση που παρέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομμάτι αυτής της ε, προσέγγισης αλληλεγγύης, όπως και για την Τινησία μέσο του ελαιολάδου ήταν σημαντικός και όπως οποιαδήποτε διμερή εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγύησεις για να εγγυηθούμε την σταθερότητα στον εσωτερική, στην εσωτερική αγορά. Ε, θεωρώ είναι ότι είναι σημαντικό σε αυτές τις ε, φάσεις να, ο μηχανισμός προειδοποίησης για πιθανή ανισορροπία στον τομέα του ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περνά και να ελέγχει τις εισεγόμενες ποσότητες. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να αποτελέσει προηγούμενο στην διαπραγματευτική διαδικασία ανάμεσα στην Ένωση και την Τινησία για τη θέσπιση μια ζώνης ελευθερού εμπορίου. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Τζουφρίντα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε στο πλευρό του λαού της Τινησίας και ως Ιταλίδα, η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει δώσει το μεγαλύτερο παράδειγμα αλληλεγγύη σε θέματα μετανάστευσης. Λέω, κύριε Επίτροπε, ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει αλληλεγγύη. Γι' αυτό και θα ήταν καλύτερο 28 χώρες της Ένωσης να συμμετείχαν στην ε, πρόταση της Κομισιόν για το μέθοδο, για τις οικονομικές της επιπτώσεις της πρότασης αυτής, ώστε να είναι πραγματική αλληλεγγύη. Αντίθετα το μέσο αυτό ε, τιμωρεί μία μόνο περιοχή, την Νότια Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα για την Ιταλία, πέρα από το ότι γεγονό είναι ιδιαίτερος και ο μοναδικός τομέας της Γεωργίας. Ε, και όλα αυτά χωρίς μελέτη τη αντικτύπου ε, ενώ οι ίδιες οι τυνησιακές ΜΚΟ μας γνωριστοποιούν ότι αυτή η συμφωνία δεν θα αρκέσει γιατί ίσως θα περιμέναν κάτι άλλο και δηλώνω λοιπόν ότι θα καταψηφίσω αυτή τη συμφωνία περιμένοντας η Κομισιόν να αναδιατυπώσει την πρότασή της για να βοηθηθεί πραγματικά η Τινησία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα ήθελα να πω εξ ότι θα υπερψηφίσω. Έχω όμως δύο δισταγμούς, δύο επιφυλάξεις. Θα υπερψηφίσω ωστόσο. Γιατί θα πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τροπολογίες ήταν καλές και πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποβούν ουσιαστικά υπέρ κάποιων διαμεσολαβητών, κάποιων ενδιαμέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τόσο πολύ προς όφελος του την ίσιου ελαιοπαραγωγού. Και γιατί? Γιατί πρόκειται για ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτό το μέτρο είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον λαό αυτό και θα πρέπει να καταδείξουμε ότι με τις ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε να υποστηρίξουμε την, την Ισία να επιστήσω όμως την προσοχή σας, γιατί τελικά θα ωφεληθούν να δείτε κυρίως οι ενδιάμεσοι. Αυτοί θα ε, πάρουν το όφελος. Ο κύριος Καπούτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με κάθε τρόπο να στηρίξει την δημοκρατισμό της Τινησίας. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομία της Τινησίας, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει εις βάρος των ελαιοπαραγωγών. Αυτή τη στιγμή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ελαιοπαραγωγικό τομέα της Ευρώπης και γι' αυτό θεωρώ πως είναι σημαντικό αύριο το Κοινοβούλιο να εκφραστεί υπέρ των διορθωτικών τροπολογιών που υπέβαλα μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Άγκρη πρώτη τροπολογία έχει στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις της πρότασης για ένα με δύο έτη. Έπειτα το λάδι θα είναι αυτό που παράγεται στην Τινησία ώστε να αποφευχθούν οι απάτες. Το πιο σημαντικό είναι το, η τέταρτη τροπολογία που προβλέπει ε, μηνιαίο έλεγχο το εισόδου των ποσοτήτων αυτών για να αποφευθεί η κατάρρευση των ευρωπαϊκών τιμών σε συγκεκριμένους μήνες ε, του χρόνου. Με αυτές τις τροπολογίες θα καταφέρουμε να βλύνουμε τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της πρότασης. Πάντως, εάν δεν υπερψηφιστούν αυτές τις τροπολογίες, θα ζητάζω να καταψηφίσω το σύνολο της πρότασης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται τη διαδικασία έτσι του Catch και στρέφουμε στην Επίτροπο Μάλστρομ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και αξιότιμοι βουλευτές. Νομίζω ότι α, η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ καλή και αυτό καταδεικνύει ότι όλοι θέλουμε να υποστηρίξουμε την Τινησία. Είναι ε, πραγματικά ευάλωτη η δημοκρατία και πραγματικά ε, πολεμάει να κρατηθεί στην επιφάνεια και ο λαός έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Ξέρουμε και τις, ε, τα χτυπήματα της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής, αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται και εμείς έχουμε καθήκον να τους βοηθήσουμε και να τους υποστηρίξουμε και η οικονομία τους έχει ε, τα πάνδυνα. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η σφαιρική και σε βάθο ζώνη ελευθερών συναλλαγών ε, έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να υποστηρίξει την οικονομία, αλλά και μια μακρότερη εταιρική σχέση και τον εκδημοκρατισμό τελικά, την διαδικασία μεταρρύθμισης. Θα συνεργαστούμε προσεκτικά με την ε, κυβέρνηση στην Τινησία να εντοπίσουμε τι προτεραιότητε, να υπάρχει αυτή η ασυμμετρία, να εξαιρούνται ε, οι τομείς που θέλουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να εισαχθούν σταδιακά. Και φυσικά θα εισακούσουμε τους φίλους μας από την Τινησία και φυσικά θα συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών στην Τινησία. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να είναι ανεκτός ο χαρακτήρας, να υπάρχει και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στην Τινησία, μιας και τόσο ευρεία η κοινωνία των πολιτών στην Τινησία. Θα υπάρχουν λοιπόν ε, μεγάλες συνέπειες ε, θετικές στο μέλλον, αλλά θα πάρει χρόνο μέχρι να τις διακρίνουμε. Θέλουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν και βραχυπρόθεσμα την Τινησία και ένα τέτοιο τρόπο είναι ο τομέας του ελαιολάδου, που είναι τόσο σημαντικός για την οικονομία του. Δεν είναι δική μα η ιδέα, ξέρετε. Είναι αξίωση, η απέτηση της Τινησίας. Θέλουμε να τους υποστηρίξουν. Θέλουν να τους υποστηρίξουμε. Πώς το κάνουμε λοιπόν αυτό. Για την νησία ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ελαιόλαδο, αυτές οι εξαγωγές. Για μας είναι μικρότερο από 2%. Φυσικά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα είναι πραγματικά περιθωριακός ο αντίκτυπος, πολύ περιορισμένος ο αντίκτυπος στην αγορά μας. Ακούω τις ανησυχίες και τους φόβους σας, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολική πολύ εξ αυτών. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και πρόκειται για ένα μέτρο για δύο και μόνο χρόνια. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένος τρόπος ε, βραχυπρόθεσμη αλλαγή προ την Τινησία. Αυτό θα καταδείξει ότι δεν περιοριζόμαστε σε όμορφα και ωραία λόγια, αλλά αναλαμβάνουμε και δράση. Και γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή πραγματικά ελπίζει ότι θα υποστηρίξει την εισηγητρία και θα υπερψήφισε την πρόταση αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Επιτροπέ. Και τώρα το λόγο έχει πάλι η εισηγητρία, κύριε Δεσέρνε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές βεβαίως στη συζήτηση αυτή και εδώ μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες, αλλά στόχος είναι ένας, να επιτύχει η την και όλος ο λαός. Δύο λόγια για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Ε, είναι σαφέ το μήνυμα του Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε απλώ συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ή εμπορική συμφωνία. Θέλουμε να αρχίσουμε μια πραγματική πολιτική εταιρική σχέση με την Τινησία. Ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει φαντασία, πραγματικά να ε, εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος μας ακούει και μας εισακούει και θα συνεχίσει και στο μέλλον. Θα πρέπει την ίση να το κάνουν κτήμα τους αυτό, να μην είναι ουρανοκατέβατες αυτές οι διαπραγματεύσεις με κάποιους εμπειρογνώμονες εντός εκτός εισαγωγικών. Ο λαός να τις κάνει. Για το δεύτερο, βεβαίω θα πρέπει να βοηθήσουμε βραχυπρόθεσμα την Τινησία, μα γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτά τα επίγοντα έκτακτα μέτρα. Και καλά κάνατε που είπατε ότι το ζητούν οι Τινήσοι. Δεν το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξύπνησε μια ωραία μέρα και να πει τι να κάνουμε σήμερα λοιπόν. Η Τινησία το ζήτησε. Και θα πρέπει να το καταλάβουν και να το ακούσουν όλοι οι συνάδελφοι. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα εδώ αλλά και ανακρίβειες για αυτά τα θέματα. Δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του συνολικού όγκου εισαγωγών ελαιολάδου από την Τινησία. Καμία, η παραμικρή. Ε, ο συνολικός όγκος θα παραμείνει ακριβώς ο ίδιος. Επιπλέον, λαμβάνουμε όλες τις προφυλάξεις. Εάν οι τροπολογίες που εμείς υποβάλαμε στην ε, Επιτροπή ψηφιστούν αύριο, γιατί ψηφίστηκαν στην Επιτροπή, μετά από ένα χρόνο θα γίνει ακριβής αξιολόγηση και αν υπάρχουν προβλήματα ανισορροπίας που σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα προκύψουν, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μέτρα αντισταθμιστικά. Ε, ζητώ λοιπόν και από όλους τους συναδέλφους να επιδείξουν ε, αλληλεγγύη, να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Οι τινήσοι περιμένουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα αύριο από εμά και ας είμαστε στο ραντεβού. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κοινή συζήτηση ολοκληρώνεται εδώ. Έχω λάβει ένα ψήφισμα για ε, να ολοκληρωθεί και